Κρίνεται. Ήμκο 14 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 25. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Ήμκο 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Για την ΙΜΚΟ 15. Beendet. Also. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 26 πέρα, 26 κατά. Να το πάλι έκλεισα. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Wir sind dann schon bei IMCO 18. Και έχουμε φτάσει στις 18 της IMCO. Υπέρ. για τη 18, ΙΜΚΟ 18. Αναφέρεται ότι είναι ταυτόσημη. Η κυρία Γκέρλινγκ ε, απέσυρε την τροπολογία της, η ΙΜΚΟ όμως δεν την απέσυρε, άρα την ψηφίζουμε. ΙΜΚΟ 18, υπέρ. Κατά. Εντάξει, οκ. Το κατάλαβα, το πιασα το νόημα. Απορρίπτεται. Κανείς δεν είναι υπέρ. Τροπολογία 39, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 11. Σε τμήματα. ο εισηγητής απέστειλε την τροπολογία, αλλά οι υπόλοιποι ε, την επανακατέθεσαν. Άρα, τροπολογία λοιπόν 11 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Να το αλλάξουμε ωραία για το δεύτερο τμήμα. Beendet. Πέρας ψηφοφορίας. Σε αυτό είχα πει, απορρίπτεται. Η 37 του Bill Newton υπέρ. Κατά. Έχετε δίκιο να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της 37. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Εντάξει. Για το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε στην 29. Σλούτερ, Άικαουτ. Υπέρ. Για την 29. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ταυτόσιμες τώρα η 10, η 30 και η 33. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 34. Α, καταπληκτή. Μάλιστα. Ωραία, καταπληκτή. Άρα τώρα είναι κάπως περίπλοκα τα πράγματα να δούμε τι καταπίπτει και περνάμε λοιπόν στην 35 τροπολογία 35 Βέσλοντ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάλι, πάλι έλεγχο. Εντάξει, ας το ξαναλέγξουμε. Για την 35. Abstimmung beendet. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εμικο 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εμικο 23 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα για την, στην ΙΜΚΟ 13. ΙΜΚΟ 13 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Στις ιτολογικές σκέψεις, ΙΜΚΟ 1, υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Α, α ναι, καταπίπτει 14. Η 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 16. Ας περνάμε στην Ίμκο 4 στο δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε στην τροπολογία 2 και ΙΜΚΟ 6. Είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο εισηγητής θέλει να ψηφίσουμε για το αρχικό κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο. Ποιος είναι υπέρ. Έχουμε δύο τμήματα. Δύο ψηφοφορίες λοιπόν. Το πρώτο τμήμα έχει να κάνει με τη λέξη household και το δεύτερο έχει να κάνει με τη λέξη laundry. Ο σας παρακαλώ, το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με τον τίτλο του όλου κανονισμού. Προτείνω λοιπόν, μολονότι έχουμε αλλάξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή μας, υπάρχουν πολλά στάδια ακόμα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι σε κάθε φάση θα προσαρμόζεται ο τίτλος του κανονισμού προκειμένου να αντικατοπτρίζει τελικά και το περιεχόμενο του κανονισμού. Αφού ζητήσετε να το ψηφίσουμε, μπορούμε να το ψηφίσουμε. Όποιοι θέλουν να ψηφίσουν κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν καταρχά τη λέξη household. Στον τίτλο υπέρ. Όχι, πρόεδρε. Der Berichterstatter hat seinen Antrag zurückgezogen. Der Rapporteur no longer wants us to vote on it, right? Also, der Berichterstatter will nicht mehr, dass wir ab. Ο εισηγητής δεν θέλει να ψηφίσουμε λοιπόν. Κύριε Νιούτον Ντάν, σας παρακαλώ, πείτε μας τι ψηφίζουμε. Πρόεδρε, στην ψηφοφορία αυτή έχουμε τροποποιήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο γενικός τίτλος. Θα μπορούσαμε να τον αλλάξουμε τώρα, αλλά απομένουν ακόμα πολλά στάδια εξέταση από το Συμβούλιο κτλ. Προτείνω λοιπόν να αφήσουμε τον τίτλο αυτή τη στιγμή ως έχει, να μην ψηφίσουμε δηλαδή τώρα και κάποια στιγμή αυτόματα αργότερα η γραμματεία, όταν θα γνωρίζουμε την τελική μορφή του κανονισμού, θα αλλάξει και τον τίτλο. Άρα δεν ψηφίζουμε. Ωραία, λοιπόν, αυτόματη προσαρμογή, καμία ψήφος λοιπόν στην παρούσα φάση. Yeah. Yes. Dann sind wir bei der... Και έχουμε περάσει λοιπόν πλέον στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. παρακαλώ. ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. 51 ψήφοι υπέρ, 8 κατά, 1 αποχή. Και τώρα για το νομοθετικό ψήφισμα, έναξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Μα λείπουν κάποιοι ψήφοι. Ωραία. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. 48 υπέρ, 8 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας για την μείωση των φωσφορικών ενώσεων στο περιβάλλον και στα ύδατα. Στο 11 τώρα τη ημερήσια διάταξης. Συνολική προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών αερίων που επιδρούν στο κλίμα, εκτός του διοξιδίου του άνθρακα. Σχέδιο ψηφίσματος μετά από μια προφορική ερώτηση του Ρίσαρτ Ζέιμπερ και του Θεόδωρου Σκυλακάκη. Έχουμε τον κατάλογο ψηφοφοριών. Η 7 της κυρίας Πλάμπ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 5B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 8. Άικαουτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε για την 8. Abstimmung beendet. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η έντεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η δώδεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στις αντιλογικές σκέψεις. Τραπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 3 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, έναξη ψηφοφορίας. Τέλος. 57 η ψήφη υπέρ, μία η κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στους συζητητές ε, Ζέμπερ και Σκυλακάκη. είδατε που πάνε τα πράγματα καλά ακόμα και αν δεν ανήκετε στην ίδια ομάδα. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι ψηφοφορίε. Σα ευχαριστώ για τη συμμετοχή σα και πάμε στο σημείο 12. Δεν έχει φτάσει λοιπόν ο εισηγητή ακόμη, γι' αυτό θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ah. όχι, θα κοιτάξουμε το θέμα αυτό. Θα περάσουμε στους κοιόδη συζητητές όμως. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού της Οικονομικής Πολιτικής. Ο κύριος Ρεβελίνη καταφτάνει. Να προτείνω λοιπόν να παρακαλέσουμε τους κοιόδης συζητητές. Έχουμε τον Κρήτον Αρσένη και του δίνω το λόγο κατευθείαν για το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, παρακαλώ να συνεχίσουν τη συζήτηση έξω, για να έχουμε λίγη ησυχία στην αίθουσα. Να έχουμε λίγη ησυχία να ακούμε τι λέμε τέλος πάντων. Ωραία. Καλύτερα. Κρήτον. Έχει το λόγο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Thank you very much, Mr. President. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με πολύ καλά σημεία. Συζητάμε σε πάρα πολλές χώρες όπως και στη δικιά μου που διανύουν μια πολύ σημαντική οικονομική κρίση την κατάσταση αυτή που ουσιαστικά απειλεί τα όσα πετύχαμε στην Ευρώπη τα τελευταία 60 χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο, θα πρέπει να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε τις τράπεζές μας, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε την οικονομική ανάπτυξη παντού στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε σε θέση να, να, είμαστε σε θέση να δανειζόμαστε με φυσιολογικούς όρους, με λογικά επιτόκια. Όλα αυτά έχουν σχέση και με τα ζητήματα που μας απασχολούν στη δική μας την Επιτροπή. Συζητάμε σε συγκεκριμένη έκθεση το ζήτημα του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Βλέπουμε πολλές φορές ότι ε, δεν υπάρχει κάποια νομιμότητα στον τρόπο που σχεδιάζεται η οικονομική πολιτική και θα πρέπει να εμπλέκεται περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με τα όσα λέει ο συγητής, πιστεύω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε κάποια πράγματα ακόμα. Δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντική πτυχή στην αξιολόγηση που προτείνεται εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής και στην επίτευξη των οικονομικών στόχων να έχουμε κατά νου και το περιβάλλον. Έχουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020, έχουμε μια έκθεση που έχει να κάνει με την απασχόληση και μια έκθεση η οποία έχει ένα μακροοικονομικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει όμως καμία έκθεση, καμία αναφορά που να έχει να κάνει με το περιβάλλον. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον, το γνωρίζουμε αυτό στη δική μας Επιτροπή, πόσο σημαντικό είναι για την ε, ήπειρό μας, για την ανταγωνιστικότητά μας. Έχουμε πάρα πολλές χώρες οι οποίες κάνουν πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις, όπως η Κίνα. Αν δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε πέρα από τους οικονομικούς μας στόχους και τους περιβαλλοντικούς στόχους, τότε θα καταφέρουμε να πετύχουμε ούτε τους υπόλοιπους στόχους που προβλέπονται στην ε, διαδικασία της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και ένα τέταρτο παράρτημα το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ο κύριο Γκερμπραντή για τους φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον Κρήτον Αρσένη για την παρέμβασή του, τη συμβολή του. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε. Διάβασα και είδα τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ασχολείται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και πιστεύω ότι πρέπει και εμείς να εργαστούμε πάρα πολύ σοβαρά. Η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε τον πλανήτη μας, αλλά ακόμα και για να προδεύσουμε οικονομικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και εμείς να μπορούμε να εμπλακούμε στο ζήτημα της βιωσιμότητας με τον τρόπο που ασχολείται και η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα οικονομικά ζητήματα. Επομένως θεωρώ ότι θα πρέπει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να εστιαστούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα στο ζήτημα της βιωσιμότητας και πιστεύω ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να σημειώσουμε μια κάποια πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη αυτής της βιώσιμης κοινωνίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης το οποίο έχει υποβάλει, για την παρούσα μορφή τουλάχιστον που έχει. Ξέρω ότι ο το μέγεθο που μπορούσε να έχει το έγγραφό ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο, θα μπορούσα εγώ να υποβάλω μια-δυο τροπολογίε για να κάνω το έγγραφο ακόμα πιο ε, ισχυρό. Θα ήθελα να αναφερθούμε περισσότερο στην, ε, στον ενεργειακό εφοδιασμό στην επάρκεια όσον αφορά τους φυσικούς πόρους. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Βλέπουμε ότι οι τιμές πολλών πόρων αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι αυξάνονται πάρα πολύ σημαντικά οι τιμές των τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να είμαστε οικονομικά αποδοτικοί με τους πόρους αυτούς. Θα ήθελα να αφαιρθώ επίσης στην ενεργειακή επάρκεια, συνεργειακή ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με τη χρήση την ενεργειακή που κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν και ως προς αυτό να υποβάλω κάποιες προτάσεις και ελπίζω πραγματικά ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής να συμφωνήσει με τις προτάσεις αυτές που θα κάνουμε εμείς για την βιωσιμότητα. Γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο σε οικονομικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε κύριε Μπράντε και ο εισηγητής μας έχει καταφτάσει πλέον. Να του δώσω λοιπόν κατευθείαν το λόγο κύριε Ριβελίνη για την έκθεσή σας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη, ήμουνα προεδρεύων στην αντιπροσωπεία Ευρώπη-Κίνα, γι' αυτό καθυστέρησα. Τώρα, μια πρόταση για την Επιτροπή ε, εδώ. Ε, ε, έχουμε και την Επιτροπή επί της Οψίας, στην Οικονομική. Κοιτάξτε να δείτε. Να ξεκινήσω τώρα. Καταρχήν, υπογραμμίζεται το θέμα της αποτελεσματικότητας των ε, πόρων και των ενεργειακών πόρων είναι πολύ σημαντικά για την βιώσιμη ανάπτυξη και για τον αγώνα κατά των κλιματολογικών αλλαγών. Μέσο και, και μακροπρόθεσμα είναι σημαντικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα. Αποτελούν σημεία κλειδιά. Μετά έχουμε εκτιμήσεις που γίνανε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πετύχουμε παρά το στόχο ε, των 20% και ότι τα σχέδια των κρατών μελών κινδυνεύουν να μην πετύχουν το στόχο, αυτό καθ' αυτό που ανέφερα, το 20% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, όπως αυτό καθιερώθηκε στην ε, στρατηγική του 2020. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν ε, απώλειες όσον αφορά την ανάπτυξη άρα ε, δεν θα δημιουργηθούν θέσεις ε, απασχόλησης. Επίσης αναφέρεται ότι υπάρχουν δυνατότητες σημαντικές ε, στα θέματα καταναλώση και κυρίως σε τομείς όπου έχουμε, που είναι ενεργοβόροι όσον αφορά το θέμα αυτό, οικοδομικός, κατασκευαστικός και μεταφορές και βιομηχανία. Επίσης, υπάρχει το νέο σχέδιο, αυτό το 2011, για την ενεργειακή απόδοση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το Μάρτι του 2011 και συνιστά όλα αυτά πρόσθετες, να ληφθούν πρόσθετα μέτρα και πιο αυστηρά μάλιστα. Πέμπτον, η Επιτροπή κάνει μια έκκληση και προτείνει ήδη από τώρα ε, περιοριστικούς δεσμευτικούς στόχους ε, στα κράτη-μέλη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και αυτό λαμβάνοντα υπόψη φυσικά τι διαφορετικέ διαφορετικές καταστάσει που έχουμε στι χώρε μέλη. Λαμβάνοντα υπόψη την οικονομική του απόδοση και τα μέτρα που έχουν ήδη Έκτον, υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για συντονισμό τη οικονομική πολιτική θα πρέπει να διαγράφεται στο εξή πλαίσιο όπου θα έχουμε μια, ένα πνεύμα μετάβαση σε μια οικονομία που είναι βιώσιμη και η οποία σέβεται το περιβάλλον. Και έβδομη πρόταση, νήξη, είναι ότι κάνει έκκληση η Επιτροπή, ε, καλείται μάλλον Επιτροπή, σε κάθε ετήσια επισκόπηση της ανάψυκτης να κάνει μια έκθεση όπου αναφέρει τους δείκτες που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντικο-οικονομική λογιστική. Αυτές ήταν λοιπόν ε, οι προτάσεις με την γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ κύριε Λιβελίνη για το σχέδιο ψηφίσματο αυτό. όντω, η Επιτροπή μας θα πρέπει να προσέξει προκειμένου να μην είναι μόνο οικονομικές οι σκέψει που θα επικρατήσουν, αλλά και οικολογικές ε, ανησυχίε σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής και του προπολογισμού στα κράτη-μέλη. Και ψηφίσαμε και μια νομοθεσία στο Στρασβούργα τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς. Ήμουν και συγκητής σε ό,τι αφορά τα έξοδα, τις δαπάνες ετησίως για περιβαλλοντικά μέτρα, ενεργειακή αποδοτικότητα, προστασία των υδάτων, ε, περιβαλλοντικά μέτρα γενικώ. Είναι σημαντικό στο ευρωπαϊκό εξάμεινο να ληφθούν υπόψη και οι πτυχές αυτές. Οι σκιώτες μίλησαν ήδη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι στην αίθουσα. Ως εκ τούτου να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το σχέδιο αυτό. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 20 Ιουνίου ώρα 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην αντιπροσωπεία με την Κίνα. Γιατί και αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο θέμα να πείτε στους Κινέζους τι κάνουμε εδώ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν κάνει κάτι παρόμοιο και η Κίνα. μου κύριε Πρόεδρε, σίγουρα θα πρέπει να κατα... κάνουμε τους Κινέζους να καταλάβουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, αλλά και εμείς, και εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο σαφείς ε, όσον αφορά τη σχέση μας και την εικόνα που για την Κίνα. Ευχαριστώ. Ναι, για την προστασία του κλίματος ε, η Ευρώπη έχει πετύχει συγκεκριμένα γεγονότα με το ενεργειακό πακέτο για την ε, προστασία του κλίματος. Παρακαλούμε με ενδιαφέρον τις κινήσεις της Κίνας και την χρειαζόμαστε την Κίνα κυρίως σε ό,τι αφορά την αγορά για την ανταλλαγή, την εμπορία ρήπων. Και θα πρέπει να κατανοήσουν αυτό το σύστημα εμπορίας ρήπων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές και τις μεταφορές και τις ε, ναυτιλιακές μεταφορές. Στην επόμενη συνεδρίαση θα καλέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αναφέρει ποιες είναι οι δυσκολίες και με την Κίνα σε ό,τι αφορά τις ε, αεροπορικές μεταφορές και τη συμπερίληψη κινέζικων αερογραμμών στο σύστημα εμπορίας ρήπων από το 2012, από του χρόνου δηλαδή. Εδώ δεν θα πρέπει να απειλούμε με την πολιτική μας, αλλά να συνεργαζόμαστε, να καταρτήσουμε μια πολιτική συνεργασίας. Και νομίζω ότι και αυτή την γραμμή θα ακολουθήσει και την αντιπροσωπεία μας. Μίλησα λίγο παραπάνω ε, γιατί για το επόμενο θέμα, για την μη αμοιβόμενη δωρεά αίματος, χρειαζόμαστε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον όμως έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να περιμένουμε λοιπόν, δύο 2-3 λεπτά μέχρι να καταφτάσει η εκπρόσωπο της ευρωπαϊκή επιτροπή Αν κάποιος από την Επιτροπή θέλει να κάνει κάποια παρουσίαση, πολύ ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω από την ε, συνάντηση των συντονιστών τα εξή. Θα καταρτήσουμε δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας για την ε, αξιολόγηση του προγράμματος ε, δράσης για το περιβάλλον και για την προετοιμασία ενός έβδομου προγράμματος δράσης. Το άλλο θέμα είναι η βιοποικιλότητα και η σχετική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό το θέμα θα υπάρξει, θα γίνει μια έκθεση. Και στη συνέχεια έχουμε δύο αντιπροσωπείες στις αρχές Σεπτεμβρίου, μία για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος στην Κομπεχάγη και άλλη μία για το ECDC, για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης ε, Νόσων στην ε, Στοκχόλμη. Να σας πω ότι το ΕΛΚ και η πράσινη... Ε, πρέπει να ορίσουν υποψήφιους για την αντιπροσωπεία στην Στοκχόλμη. Στην ε, Ολομέλεια θα καταθέσουμε ένα προφορικό ερώτημα με το ψήφισμα για την ε, επόμενη παγκόσμια συνάντηση σύνοδο στην Βραζιλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ορίσει την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλλει από πλευράς του με ένα ψήφισμα. Θα πάμε επίσης στην EMA στο Λονδίνο την παράλληλη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη. Αναζήτησε λοιπόν ένα νέο εκτελεστικό διευθυντή, τον οποίο και βρήκε εδώ μεταξύ, τον ε, όρισε Και ο νέος διευθυντής λοιπόν ονομάζεται Γκίντο Ράζι από την Ιταλία. Ο οποίος ήταν εκεί επικεφαλής ε, της ιατρικής υπηρεσίας και από 13 Ιουλίου το, μάλλον στις 13 Ιουλίου το απόγευμα θα διοργανωθεί η ακρόαση να ακούσουμε πώς φαντάζεται ότι θα δημορφωθεί το μέλλον της υπηρεσίας. Και μετά θα ψηφίσουμε, μετά την ολοκλήρωση της ε, ακρόασης. Όπως σας είπα, μιλήσαμε για τις ε, δυσκολίες σε ό,τι αφορά το σύστημα εμπορίας τύπων ε, για τις αερομεταφορές. Η Κίνα μας απείλησε πραγματικά και είπαμε σήμερα το πρωί στους συντονιστές ότι κάποιες ε, ότι είναι Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί ότι θέλει, αλλά από το 2009 υπάρχει ένας νόμος, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε πλέον. Άρα, ως ε, ε, Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή στι διαπραγματεύσει με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τις αερογραμμές αλλά και τι διαπραγματεύσει με την Κίνα. Να αναφέρω και ένα άλλο θέμα παρόλα αυτά. Φυσικά απευθύνομαι σε όσους βρίσκονται εδώ στην αίθουσα. Η Επιτροπή αυτή αποφάσισε τη διοργάνωση κάποιων ακροάσεων. Αλλά η συμμετοχή στις ακροάσεις είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητική. Και έχουμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα μία ακρόαση. Α, την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, Για την προστασία του περιβάλλοντος στην Βαλτική θάλασσα. καλό θα ήταν να μην, να μην συμμετέχουμε μόνο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αλλά και στις ε, ακροάσεις που διοργανώνονται. Έγινε επίσης και μία αναφορά για την ε, κακή διατροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί ασφαλώς ένα μεγάλο θέμα αυτό, η κακή διατροφή. Θα δούμε λοιπόν αν θα ασχοληθεί επισήμως η Επιτροπή με το θέμα αυτό. Να παρακαλέσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει εδώ στην Επιτροπή μας για να μας μιλήσει για το θέμα της επιβάρυνσης ε, με ακτινοβολία λόγω των κινητών τηλεφώνων και την ενδεχόμενη, ε, τον ενδεχόμενο κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου από την ακτινοβολία στην επόμενη συνεδρίασή μας. Επίσης, συζητήσαμε τι θα κάνουμε με την ε, αποτυχημένη προσπάθεια που έγινε για τα καινοτόμα τρόφιμα. Θα στείλουμε μία επιστολή στον Επιτροπό Ντάλι για να, να ρωτήσουμε πότε θα υποβάλει νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τα νέα τρόφιμα αυτά συγκέντρωσαν μεν ομόφωνη υποστήριξη, αλλά τελικά ήταν υπερβαλλικά αμφιλεγόμενο το θέμα της κλωνοποίησης και στο, στην Ολομέλεια η Επιτροπή είπε ότι θα υπάρξουν δύο πρωτοβουλίες. Καταρχάς μία για τα καινοτόμα τρόφιμα και άλλη μία για την κλωνοποίηση. Αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει στο εγγύς μέλλον. Γιατί εισάγονται πολλά υλικά και υπάρχει και το θέμα ε, των απογόνων των κλωνοποιημένων ζώων. Μάλιστα. Μίλησα λοιπόν. Ο συνάδελφος Σνέλχαρτ ήθελε να κάνει μια παρατήρηση και έχει καταφτάσει ήδη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο θέμα. Ναι, ο κ. για το τελευταίο αυτό ζήτημα θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξή στην επιστολή να γίνει αναφορά και στο εξή στοιχείο. Παρά το γεγονός ότι όλοι συμφωνούμε για τα νέα καινοτόμα τρόφιμα, ε, θα θέλαμε να υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν η πρόταση αυτή και να υπερψηφιστεί. Γιατί δεν έχω καμία όρεξη να ξαναζήσω τέτοιες λαϊκιστικές ε, ενέργειες. Πολύ σωστό αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι και οι δύο προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν γρήγορα, αλλά αν δεν το καταφέρουμε αυτό, ας καταφέρουμε τουλάχιστον να έχουμε στα καινοτόμα τρόφιμα μία πρόταση, να ρυθμιστεί νομοθετικά το συντομότερο δυνατόν, γιατί βλέπουμε συχνά και σε θέματα νανοτεχνολογίας, ε, μεγάλες εξελίξεις. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε γρήγορα για την κλωνοποίηση των ζώων. Πιστεύω, συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να ελέγξουμε στα σοβαρά και πάλι τη στάση μας. Τον τελευταίο καιρό έχω ενημερωθεί κάπως και ξέρετε ζούμε ίσως όχι απόλυτα με στην πραγματικότητα. Μας ξεπερνούν οι εξελίξεις. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να παρακολουθούμε με τις ε, νομοθετικές ε, διατάξεις μας, τις εξελίξεις. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν μια συζήτηση στο ιστορικό της ομάδας για να αναδιαμορφώσουμε ενδεχομένω τη θέση μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Το συζητήσαμε το θέμα και η κατήκα Λίοταρτ, ε, η συγγήτρια, επιθυμούσε να καταρτήσει έκθεση πρωτοβουλία, απευθύνοντα έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάθεση νομοθετική πρόταση. Έχουμε το δικαίωμα αυτό με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνα. Άλλε ε, επιτροπές ε, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το άρθρο 225 της συνθήκης της Λισαβόνα. Ήταν θέμα διαδικαστικό. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να Υποβάλλει το συντομότερο δυνατόν πρόταση και να αναλάβει και πρωτοβουλία. Απλά, λέει ο κ. Σνέλχαρτ, πιστεύω ότι σε θέματα κλωνοποίησης θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την θέση μας. Ιδάλλως, μπορεί να μην ε, καταλήξουμε και πάλι σε κάποιο αποτέλεσμα και θα μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις. Δεν ξέρω ποια θα είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει να συμβάλλει και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μετά την ενημέρωση του τελευταίου καιρού, θεωρώ ότι ίσως να είμαστε κάπως υπερβολικά αυστηροί. Ναι, κοιτάξτε, ε, το παιχνίδι έχει ξαναρχίσει μετά την αποτυχημένη προσπάθεια την τελευταία. Θα πρέπει να, κατα... να υποβάλει νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά θα την ελέγξουμε εμείς, έχουμε και το Συμβούλιο, ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη με τα 27 κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον θα υπάρξει μια δεύτερη αποτυχία ή μήπως στην δεύτερη προσπάθεια καταφέρουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό για να υπάρξει μια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ως τώρα δεν έχουμε ρύθμιση, κάνει ό,τι θέλει η αγορά και δημιουργεί μια κατάσταση de facto. Νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε στο θέμα αυτό και μετά τις θερινές διακοπές θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ωραία λοιπόν. Άρα περνάω στο θέμα 13 αυτή τη στιγμή για το θέμα της ε, δωρεάς αίματος, τις διαδικασίες, τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται από πλευράς Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ε, έμειναν εδώ πέρα όλοι οι δωρητές αίματος. Είναι πάρα πολύ λίγοι όμως τον αριθμό. Θα έπρεπε να είναι πιο πολύ Ιδιαίτερα στην επιδημία ΙΧΕΚ έγινε έκκληση στη χώρα μου από τα νοσοκομεία για δωρεά αίματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και εγώ όσο πιο συχνά μπορώ δίνω αίμα. Να μας αναφέρει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρισκόμαστε, πώς έχει κατάσταση. Έχουμε μαζί μας ο κ από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και ο Στέφαν Φαντεσπίγκελ, επικεφαλής για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης. Δύο αρμόδιους έχουμε λοιπόν μαζί μας σήμερα. Σας παρακαλώ κάντε μας μια εισαγωγή στο θέμα. Yes, thank you, Mr. Chairman. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αντιμάνω ονομάζομαι και είμαι επικεφαλής της μονάδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια για το αίμα, τις μεταγγίσεις αίματος, καθώς επίσης και τη δωρεά οργάνων. Ο συναδελφός μου εδώ σήμερα δεν είναι δημοσιογράφος όπως ακούστηκε, είναι ο συναδελφός μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Την κατάλληλη στιγμή λοιπόν πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην Επιτροπή σας γιατί ε, χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα δωρεάς αίματος οργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και γίνανε διάφορες δραστηριότητες πρόθεσης και προβολής ε, της δραστηριότητας αυτής. Επίσης όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και κάποιους μήνες έχει ε, δημοσιοποιήσει μία έκθεση για την εθελοντική και μία αμοιβόμενη δωρεά αίματος. Και είναι η έκθεση την οποία θα σας παρουσιάσουμε σύντομα. Και στη συνέχεια θα θέλαμε να πούμε και κάποια πράγματα για τα μελλοντικά βήματα στον τομέα αυτό. Ξεκινάω λοιπόν αναφερόμενος στο τι εννοούμε όταν λέμε εθελοντική και μη αμοιβόμενη δωρεά αίματος. Ουσιαστικά είναι μια γενικά αποδεκτή αρχή ότι η δωρεά αίματος θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και όχι στην αρχή της, του οικονομικού κέρδους Υπάρχει μία, ένας ορισμός από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον οποίο έχουμε συμπεριλάβει και στην έκθεση αυτή. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στην δωρεά αίματος, η οποία γίνεται εθελούσια, χωρίς να υπάρχει κάποια χρηματική αποζημίωση ή αποζημίωση αμοιβή σε είδος. Δεν χρησιμοποιείται δηλαδή κάποιο άλλο μέσο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των χρημάτων. Σαφώς θα μπορεί η δωρεά αίματος να συνοδεύεται με κάποια μικρά δώρα ή με προσφορά αναψυκτικών ή με την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου κτλ. Και το έχουμε μελετήσει αυτό και στην έκθεσή μας. Δηλαδή τι είδους διευκολύνσεις τι είδους κίνητρα πολλές φορές ε, δίνονται προς τους δότες προκειμένου να ε, δώσουν αίμα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε επίσης και το νομικό πλαίσιο. Η αρχή της εθελοντική και μη αμοιβόμενης δωρεάς αίματος δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, η οδηγία λέει ότι τα κράτη-μέλη θα θα προχωρήσουν στα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθελοντική και μη αμοιβόμενη αιμοδοσία. Σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζεται ως μια νομικά δεσμευτικά αρχή. Και στη συνέχεια βέβαια υπάρχει και αυτή η υποχρέωση υποβολής αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των οποίων δημοσιεύονται οι εκθέσεις αυτές. Η πρώτη έκθεση δημοσιοποιήθηκε το 2006 και τη ξέρετε ότι η οδηγία είναι του 2002. Στην πρώτη μας λοιπόν έκθεση είχαμε εντοπίσει την ανάγκη να γίνει μια ανταλλαγή εμπειριών και βελτίστων πρακτικών. Έκτοτε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια σειρά από μελέτες και παρουσιάσαμε δύο από τις μελέτες αυτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρώτη μελέτη είναι μία μελέτη που φέρει τον τίτλο Domain Project. Ουσιαστικά καταφέραμε να πετύχουμε μία συλλογή βέλτιστων πρακτικών που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των δωρητών, δηλαδή όλη η διαδικασία αυτή που έχει να κάνει με την προσέλκυση των αιμοδοτών και όλη η διαδικασία της ε, προώθησης και της προβολής της αιμοδοσίας προκειμένου να καταφέρουμε να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή όλα αυτά τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε, φυλάδια, ενημερωτικά κτλ. προκειμένου να καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερους αιμοδότες. Και στη συνέχεια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε τους υφιστάμενους αιμοδότες. Τα άτομα δηλαδή τα οποία ήρθαν και δώσαν αίμα μια πρώτη φορά να συνεχίσουν να πράττουν αναλόγους και στο μέλλον. Αυτό Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να καλύψουμε στη μελέτη αυτή που είχε να κάνει με τη διαχείριση των αιμοδοτών. Είχαμε όμως και μια δεύτερη έκθεση που είχε να κάνει με την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση του αίματος, Optimal Blood Use. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην δεύτερη αυτή έκθεση, την οποία μόλις δημοσιεύσαμε. αναβλήθηκε η δημοσιοποίησή της προκειμένου να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε και τα πορίσματα των ε, μελετών αυτών στις οποίες αναφέρθηκα. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε κατά ποιον τρόπο οι βέλτιστες αυτές πρακτικές αντικατοπτρίζονται στα κράτη-μέλη, πόσο ευρέως χρησιμοποιούνται, λάβαμε απαντήσεις από 27 κράτη-μέλη και από την Κροατία και την Νορβηγία. Τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους επικεντρωθήκαμε και για τους οποίους θέσαμε ερωτήσεις στα κράτη-μέλη. Καταρχάς, αν έχουν μια κάποια νομοθεσία η οποία ενθαρρύνει την εθελοντική και μια αμοιβόμενη δωρεά αίματος, ποια κίνητρα χρησιμοποιούν και ποια μέτρα προώθησης χρησιμοποιούν και στη συνέχεια πώς οργανώνουν την συλλογή και την προμήθεια. Και έχετε μία σύντομη περιγραφή στην έκθεση αυτή για κάθε έναν από τους τομείς αυτούς. Οι περισσότερες χώρες, σχεδόν όλες μάλιστα θα έλεγα, χρησιμοποιούν μια κάποια νομοθεσία, έχουν πλέον νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να προωθήσουν την ε, εθελοντική και μη αμοιβόμενη δωρεά αίματος. Και πολλές φορές προβλέπονται και κάποιες κυρώσεις. Σε 15 χώρες συγκεκριμένα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται μια σειρά κινήτρων για την πρόθεση της δωρεάς αίματος, κίνητρα τα οποία δίνονται ουσιαστικά στους δότες και ουσιαστικά τα κίνητρα αυτά τα βλέπετε και στον πίνακα που έχετε μπροστά σας. Αναψυκτικά, μικρά δώρα, αποζημίωση των δαπανών ταξιδίου, άδεια, δωρεάν υγειονομικό check-up κτλ. Επίσης προβλέπονται και στη συνέχεια κάποια μέτρα προώθησης, προβολής, που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού. Διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης, διάφορες οι μερίδες οι οποίες οργανώνονται για την ευαισθητοποίηση του κοινού, όπως για παράδειγμα η μέρα της αιμοδοσίας, διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες οργανώνται κυρίως σε εθνικό επίπεδο και έχουν ως στόχο την προσέλκυση νέων δοτών και τη διατήρηση των υφισταμένων. Πολύ συχνά επίση οι καμπάνιες αυτές, οι εκστρατείε αυτές στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως φοιτητέ, υπηρετούνται στο στρατό κτλ. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι να δούμε πώς οργανώνεται η συλλογή των δεδομένων στα κράτη-μέλη. Αυτό γίνεται κυρίως μέσω του δημοσίου φορέα, μέσω συγκεκριμένων δημοσίων κέντρων αιμοδοσίας. Στη συνέχεια να αναφερθούμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο διαδραματίζει ένα πολύ θεμελιώδη ρόλο στον τομέα αυτό και το λέω αυτό και εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δημιουργήσει ένα οργανισμό σφαιρικό που συντονίζει την έρευνα στον τομέα της αιμοδοσίας και που έχει ως στόχο επίσης και τη γενικότερη διαχείριση των αιμοδοτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στεργαζόμαστε λοιπόν εμείς πολύ στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης για το ζήτημα αυτό. Και μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μία μελέτη για να εντοπίσουμε για παράδειγμα τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την προσφορά αίματος, την προσέλκυση νέων δοτών κτλ. Τι προβλέπουμε να κάνουμε τώρα στο μέλλον. Υπάρχουν κάποιες αρμόδιες εθνικές αρχές, των οποίων ηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Έγινε μια συζήτηση της έκθεσης αυτής ε, με τους φορείς αυτούς τον ε, Μάιο λοιπόν. Εξετάσαμε επίσης και τις μελέτες που ε, δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Το συμπέρασμα της συνάντησης αυτής ήταν ότι δεν υπάρχει λόγος να εγκριθούν περαιτέρω νομοθετικές διατάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εθελοντική και μη αμοιβόμενη δωρεά αίματος. Με η υφιστάμενη νομοθεσία, οι υπάρχοντες νόμοι αντικατοπτρίζουν ε, πολύ καλά τις, τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα πρέπει να ρυθμιστεί ο τομέας της εθελοντικής και μη μιβόμενης δωρεάς αίματος. Δεν υπάρχει δηλαδή ανάγκη για περαιτέρω νομοθεσία θα είμαστε σε συνεχή μελλοντική επαφή και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τους έχουμε μάλιστα ζητήσει να υποβάλουν μία αναφορά προς τις ευρωπαϊκές εθνικές αρμόδιες αρχές για, την, για τα περαιτέρω πορίσματα που θα έχουν στις μελέτες τους. Και στα τέλη του 2013 θα έχουμε και την επόμενη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Πολύ καλή εισαγωγή αυτή που μας κάνατε και θα αποτελέσει πολύ καλή βάση για τη συζήτηση την οποία θα έχουμε. Δεν ξέρω αν ο συναδελφό σα θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι, μάλιστα. Σε αυτή τη φάση δεν θέλει να πει τίποτα. Ναι, πράγματι αναφέρετε κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Παρακολουθώ στην παλτρίδα μου και βλέπω ότι οι νέες γενιές όλο και λιγότερο ε, πάνε να δώσουν αίμα σε σχέση με τις παλαιότερες ε, γενιές. Ε, έχει εντοπιστεί αυτό το πρόβλημα, παρουσιάζεται και σε άλλες χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να παρατρύνουμε και τους νέους. Να δίνουν αίμα. Γιατί αν δεν έχουμε πλέον αίμα, θα είναι ασφαλώς τεράστιο το πρόβλημα που θα αντιμετωπίζουμε στην υγειονομική περίθλαψη. Ο κύριος Μικολάσεκ ζήτησε το λόγο. Ďakujem, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ε, η εθελοντική και μη αμοιβόμενη δωρεά αίματος είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το συζητάμε εδώ σήμερα. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την αιμοδοσία. Οι νέοι δεν διέπονται από την νοτροπία αυτή της αλτρουιστικής δωρεάς αίματος, της εθελοντικής δωρεάς αίματος. Δεν είναι τόσο εύκολα πρόθυμοι να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένη νοοτροπίας η οποία χάνεται όλο και περισσότερο και πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να σχεδιάσουν κάποιες νέες πολιτικές, κάποιες νέες ενημερωτικές εκστρατείες για να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τους νέους. Ξέρετε ότι η ανάγκη για αίμα θα υπάρχει πάντοτε, αλλά δυστυχώ βλέπουμε ότι όλο και μειώνται οι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να δώσουν αίμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν αίμα σε όλα τα εθνικά συστήματα υγεία. Υπάρχουν διάφορε προκλήσει τι οποίε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπω για παράδειγμα η πρόσφατη επιδημία στη Γερμανία. Εποφελούμε τι ευκαιρίε για να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή. και πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε δραστηριότητες που θα έχουν ως στόχο να προωθήσουν την εθελοντική δωρεά αίματος. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση για την αιμοδοσία, γιατί ε, αν ακολουθούσαμε το δρόμο αυτό θα εμπορευματοποιούσαμε τελικά την όλη διαδικασία και ουσιαστικά το αίμα θα ήταν διαθέσιμο μόνο σε αυτού που θα είχαν τα χρήματα για να το αγοράσουν. Πιστεύω ότι η αρχή τη εθελοντική δωρεά αίματο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπε πριν από λίγο ο συνάδελφός μας. Σίγουρα υπάρχουν εκστρατείε ενημέρωσης οι οποίες όμως δεν αρκούν στις χώρες μέλη που γίνονται μας είπαν ότι η νομοθεσία ήταν καλή. Σημάμαι, σημάμαι πολύ καλά. Είχαμε τότε μια συζήτηση όταν ψηφίσαμε για αυτή την οδηγία. Αλλά, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν εκστρατείες ενημέρωσης που είναι ε, δυνατές, ε, επαναλαμβανόμενες, αυτές θα πρέπει να συνεχίζονται με σωστή ενημέρωση σε όλους τους δημόσιους χώρους, πανεπιστήμια, χώρους όπου συχνάζουν οι νέοι. Ε, πραγματικά πρέπει να συμβάλλει η νεότητα σε αυτό. Ε, δε, σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα, μια κατάσταση όπου θα είναι κανείς υπερήφανος να, και να νιώθει αυτή τη γενοδορία, να δίνει αίμα. Αλλά θα θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Είμαστε σίγουροι ότι οι χώρες, στις χώρες μέλη ότι δεν υπάρχουν κάποιοι πειρασμοί για να αγοράσει κανείς ε, αίμα σε τρίτες χώρες φέρει πίνη. Υπάρχουν σωστοί έλεγχοι. Απαγορεύεται, εντάξει, αλλά οι έλεγχοι είναι αυτοί οι σωστοί, διότι είναι θέμα ασφαλείας. Ξέρετε, άμα καταλήξουμε μια μέρα ότι από τη στιγμή που αγοράζει κανείς αίμα δεν θα υπάρχει ε, ασφάλεια, δεν θα υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσει από τον δότη. Το ότι είναι δωρεάν η, δωρεά του αίματος σημαίνει ότι υπάρχει μια διαδικασία, ελέγχουμε τον δότη υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι ερυπίνοι για του οποίου απογορεύεται για διάφορους λόγους, άρα διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Αν μια μέρα υπάρξει έλλειψη φερπίν, δεν θα υπάρξει ο πειρασμό να γίνει εμπόριο πλέον με το αίμα. Και τότε θα έχουμε προβλήματα ασφαλείας όσον αφορά αυτό το θέμα. Και τώρα που μιλάμε για δωρεά να Εφισώ την, προσοχή, και απευθύνουμε στην Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Δεν είναι της ίδιας σε αυτό το θέμα. Έχουμε να κάνουμε τη δωρεά αίματος και οργάνω, φερμίν. Να πω όμω απλώ. Διότι είναι σημαντικό το θέμα. Ναι και συζητάμε με την Επιτροπή. Μήπως θα έπρεπε να υποχρεωτική να κρατάμε το αίμα του ομφαλίου λόρου και τον ίδιο τον ομφάλιο λόρο. Αυτό γίνεται σε ορισμένες ε, ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους ε, στα μευτήρια, αλλά δεν γίνεται σε μεγάλη κλίμακα. Ξέρουμε ότι το αίμα του ομφαλίου λόρου και ο ίδιος ο Φάλιος Λόρος είναι, ε, σημαντική, είναι σημαντικά για την έρευνα την ιατρική, για θεραπείες και για μελλοντικά φάρμακα. Ίσως εντάξει δεν έχει να κάνει τίποτα με το θέμα αυτό καθ' αυτό της ζωράς αίματος αλλά μήπως θα μπορούσαμε να το δούμε μελλοντικά να θίξουμε αυτό το θέμα διότι είναι θεμελιώδος να δημιουργηθεί αυτή η υπόχρωση να μην τα θεωρούμε θέματα τα οποία, ας πούμε, πράγματα τα οποία τα χάνουμε αλλά να τα ε, χρησιμοποιούμε. Συγγνώμη που λίγο έτσι βγήκα λίγο από το, το, το πνεύμα της συζήτηση, αλλά θεώρησα σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Θα έχουμε ίσως απάντηση αργότερα. Ο Κύριο Σνέλχαρτ. Ναι, μέχρι και στα γαλλικά το κατάλαβα ότι παίρνω το λόγο. Μάλιστα. Πρόεδρε, είναι ωραίο το ότι ακούμε μία έκθεση ότι λειτουργεί η νομοθεσία την οποία αποφασίσαμε. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά πιστεύω ότι αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, στην προβληματική του ΕΧΕΚ, είδαμε στη Γερμανία ότι υπάρχει γενικώ μία καθυστέρηση. Πώς έχει λοιπόν η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή βοήθειας για αίμα μεταξύ των κρατών μελών ρυθμίζεται αυτό μόνο σε κάθε κράτος μέλος ή υπάρχουν διασυνοριακές δυνατότητες και πώς αξιοποιούνται. Πόσο συχνά χρειάζεται και δεύτερη ερώτηση για αυτά που είπε η κυρία δευτερη ερωτηση για αυτό που ειπε η κυρια γκροστετ Δεν είμαι βέβαιος αν δεν συμβαίνουν ε, εισαγωγές από τρίτε χώρες. Υπάρχει κάποια επισκόπηση, μπορούμε κάτι να πούμε ή ίσως ε, επικρατεί η άποψη ότι, εν πάση περιπτώσει, σε καταστάσει εκτάκτου ανάγκη θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Αυτά τα ερωτήματα μα απασχολούν. Γιατί είδαμε ότι, για παράδειγμα, σε, σε καταστάσει εκτάκτου ανάγκη υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και πολλέ μικρέ χώρε ίσω να μην έχουν τι δυνατότητε που έχουν οι μεγάλε χώρε. Οι χώρε αυτέ είναι διατεθειμένε να βοηθήσουν ή επικρατούν τα σύνορα. Ευχαριστώ. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Αναφερθήκατε στην ανταλλαγή πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πώ διοργανώνεται ο συντονισμό αυτό όσον αφορά τα επίπεδα προμήθεια, για παράδειγμα. Ξέρετε πώ έχει προμήθεια σε κάθε χώρα, ποιε είναι οι ελλείψει, γίνονται ανταλλαγέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει κάποιο οργανισμό ο οποίο συγκεντρώνει τι πληροφορίε αυτέ και κάπω τι συντονίζει. Μπορούμε να γνωρίζουμε ότι για παράδειγμα στη Γαλλία υπάρχει ένα μεγάλο πλεόνασμα αίματος και μπορεί να προμηθεύσει ενδεχομένως και τη Γερμανία η οποία μπορεί να έχει έλλειψη. Okay. Ωραία, λοιπόν, αυτέ ήταν οι ερωτήσει ε, και τα σχόλια. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα απαντήσει. There Τέσσερις ήταν οι ερωτήσεις. Η πρώτη είχε να κάνει με τους νέους, άλλη μία είχε να κάνει με τις τρίτες χώρες. Είχαμε μία ακόμα ερώτηση για το αν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κρατών σε περίπτωση ατυχημάτων. Προτού απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις και προτού δώσω το λόγο στον εμπειρογνώμονα, θα ήθελα να πω ότι ε, τα όσα είπα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για τη διαχείριση των ε, δοτών κτλ. έχουν ως στόχο να υπάρχει μία επάρκεια στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μην ε, εμφανίζονται πολύ αυξημένες ανάγκες εισαγωγής ή εξαγωγής αίματος. Εμέσως αστικά αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι αυτή η αυτάρκεια των κρατών μελών. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε μέσω των εκστρατιών προώθηση τη αιμοδοσία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κίνδυνοι με την εξαγωγή και εισαγωγή αίματος καθότι δεν μπορεί κανεί να ελέγξει 100% ότι το αίμα αυτό προέρχεται μέσω τη μη αμοιβόμενη και θελοντική δωρεά αίματο ή αν είναι ενδεχομένω αίμα το οποίο έχει δοθεί με χρηματική αποζημίωση, με κάποια χρηματική αμοιβή. Ενδεχομένως ο Στέφαν θα μπορούσε να πει κάποια περαιτέρω πράγματα για να απαντήσουμε με καλύτερη ακρίβεια σε ερωτήσεις οι οποίες ακούστηκαν. Όπως είπαμε, στόχος της νομοθεσίας είναι να προωθηθεί η αυτάρκεια των κρατών μελών Θα πρέπει λοιπόν η μεγαλύτερη τουλάχιστον ποσότητα αίματος να προέρχεται από μια εθνική δραστηριότητα. Το αίμα δηλαδή θα πρέπει να συλλέγεται σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο κράτους μέλους. Βέβαια, ορισμένε φορέ πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιε κρίσει εκτάκτου ανάγκη και στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποθέματα αίματο από άλλε χώρε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να υπάρχει επαφή και στονισμός ανάμεσα στα κέντρα αιμοδοσίας, στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίσουμε ποια είναι η ζήτηση και ποια είναι η προμήθεια κάθε φορά και ακριβώς με τις εθνικές αυτές αρχές συνεργαζόμαστε στις συναντήσεις που διοργανώνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε φορά που διεξάγουμε μια έρευνα ή μια μελέτη. Μας ρωτήσατε αν εμφανίζονται ελλείψεις αίματος, όχι πολύ συχνά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η εθνική προμήθεια αίματος καλύπτει τις εθνικές ανάγκες, την εθνική ζήτηση. Όπως σας είπα όμως προκύπτουν κάποιες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπου πρέπει να καταφύγουμε και σε παροχή αίματος από κάποια άλλη χώρα. Ακούστηκε και το ζήτημα της ευαισθητοποίησης των νέων Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τις εθνικές αρχές οι οποίες έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν το κοινό. Όπως θα είδατε και στην ε, παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Μάνου, έχουμε εντοπίσει κάποιες συγκεκριμένε ε, ομάδες, όπως για παράδειγμα τους νέους ή πιο συγκεκριμένα τους φοιτητές ή τους ε, υπηρετούντες στο στρατό. Θέλουμε ουσιαστικά να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε ομάδες νέων οι οποίοι θα συνεχίσουν και στο μέλλον να είναι Όσον αφορά το αίμα από τον Οφάλιο λόρο, συμφωνώ με το σχόλιο το οποίο ακούστηκε. Όντω διεξάγονται αυτή τη στιγμή πολλέ συζητήσει για το ζήτημα αυτό. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος παρουσιάζει πολύ μεγάλες δυνατότητες για την ιατρική έρευνα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν εντοπιστεί όμως πάρα πολλές θεραπείες οι οποίες, θα μπορούσαν να προκύψουν. Ενδεχομένως όμω να έχουμε νέε θεραπείες χάρη στην έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Σε εθνικό επίπεδο πάντως διεξάγονται αυτή τη στιγμή συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να συντονιστεί η διαχείριση του αίματος αυτού Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα σημεία. Δεν ξέρω αν ξέχασα να απαντήσω σε κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μικολάσκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία σύντομη παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, απευθυνόμενος προς τον προελίσαντα. Να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα οποία είπε η Φρανσουάς Γκροστέτ πριν από λίγο. Μία ομάδα επισκέφθηκε ένα πολύ γνωστό Ινστιτούτο στη Λιόν της Γαλλίας και στην επίσκεψή μας αυτή, στην οποία συμμετείχα και εγώ, είδαμε ότι ε, το Ινστιτούτο αυτό είχε προχωρήσει στην ε, χρησιμοποίηση των βλαστοκυτάρων που μπορούν να προκύψουν από το αίμα του ομφαλίου λόρου. Χρησιμοποιήσουν επίσης και κάποια άλλα συστατικά του αίματος, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θεραπείες. Ε, το Ινστιτούτο πάντως αυτό, το οποίο είναι σίγουρα πρωτοποριακό, είχε ήδη αρχίσει να κάνει θεραπείες χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτό το αίμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα υποσχόμενες για το μέλλον. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση αυτή και την καταγράφη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε ότι στην Λιόν έχουμε ένα ιδιαίτερα προωθημένο κέντρο έρευνας. Θα είναι αυτό ιδιαίτερα χρήσιμο για πάρα πολλές εφαρμογές και στόχους. Μάλιστα, ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σίγουρα θα μας χρησιμεύσει αυτή η παρουσίασή σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνεδρίασή μας. 21 ε, Ιουνίου η επόμενη συνεδρίαση εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Sehr erfreulich, dass wir etwas früher sind. Äh, I gained one hour to do something in my office, which is fantastic. Fantastic for me as well. okay. <laughs> Thank you